σε σχέση με την εξέταση της πολιτικής μας όσον αφορά το μέλλον, την, το άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ελήφθησαν έξι προτάσεις ψηφίσματος για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψήφιση θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έδωσαν μήνυμα ότι ήθελαν να παρέμβουν και φαντάζομαι ότι αναφέρονται στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης όταν θα έρθει η ώρα για το Catch the Eye και έτσι θα, έχουν, ε, θα ληφθούν υπόψη και θα σημειωθούν για να παρέμβουν αλλά αντίστοιχα το επόμενο σημείο είναι οι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή όσον αφορά την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε. Μου ανέφεραν και πάλι ότι πιέζει ιδιαίτερα ο χρόνο και γι' αυτό θα ήθελα να σα απευθύνω έκκληση σε όλου σα να προσαρμόσετε τι παρεμβάσει σα. Ακόμα και προ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να απευθύνω αυτή την έκκληση. Να είναι συντομότατη ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα θέματα τη ημερήσια διάταξη έγκαιρα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα παρέμβει ο κύριος Νέμετ, εξ ονόματος του Συμβουλίου πάλι, για τη δήλωση που έχει να δώσει. Έχετε τον λόγο κύριε Νέμετ, παρακαλώ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση απόλυτα δεσμεύεται για την ε, τέταρτη αυτή διάσκεψη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που θα διεξαρθεί στην Ισταμπούλ από τις 29 μέχρι 30 Μαΐου του 2011 και αυτή η διάσκεψη θα είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία να διευρυνθεί η υποστήριξη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το Συμβούλιο πολύ πρόσφατα υιοθέτησε συμπεράσματα για την χρήση ως κατευθυντήριων γραμμών ως προσανατολισμών από πράσινη Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης είναι ανάγκη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να προσπαθήσουμε να τις βοηθήσουμε και γι' αυτό συνεχίζουμε να ε, είμαστε δεσμευμένοι υπέρ της αηφόρου ανάπτυξης ε, όλων αυτών των ε, χωρών που έχουν την ανάγκη βοήθειας και είναι οι φτωχότερες στη διεθνή κοινότητα και χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη, τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα τους εξωτερικές θεομηνίες, προκλήσεις και ασθένειες, πανδημίες και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε μέτρα που μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη αξία, ιδιαίτερα όσον αφορά αυτέ τι ανάγκε που έχουν και που πρέπει να αντανακλούν τα μαθήματα που έχουμε συναγάγει από το πρόγραμμα δράση των Βρυξελών, διατηρώντα σε συνεκτικότητα και ε, συνάφεια του συγκεκριμένου στόχου υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Και μια νέα εταιρική σχέση για αυτέ τι χώρε από πλευρά μα με τα εύθετα μέτρα σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα. Ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη ότι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η έκβαση αυτή τη ε, Συνόδου της Ισταμπούλ θα πρέπει τρεις κύριους στόχους να αντιμετωπίσει. Να αντιμετωπιστεί η ιδιαίτερα ευάλωτη αυτή ε, πλευρά που έχουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Δεύτερον, να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αηφορία στην ανάπτυξη των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών. Τρίτον, να προαχθεί η αηφορία στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών. Αυτοί οι στόχοι θα, θα συνεχίσουν να εμπνέουν συζητήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκαταρκτικά πριν από την Σύνοδο αλλά και κατά την Σύνοδο αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ρόλο πάντα προπομπού ε, στην διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη αυτών των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών και ήταν ο μεγαλύτερο χορηγό. Ήταν ο πιο ε, ισχυρό ε, και αποτελεσματικός εταίρος με τη συνδρομή που έδινε και για την πρόσβαση στην αγορά, προσπελασιμότητα στην αγορά, κανόνε προέλευση και σημειώθηκε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και για την συνεκτικότητα της πολιτικής υπέρ της ανάπτυξης. Κάποιες από αυτές τις χώρες έχουν σημειώσει θετική οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο κατά τα τελευταία χρόνια. Όμως αναγνωρίζουμε ότι συνολικά η πρόοδος αυτή ήταν άνηση και πολλή δουλειά πρέπει ακόμα να γίνει. Κυρίως στην υποσαχάρια συμβρινή Αφρική και στις χώρες που βρίσκονται και αντιμετωπίζουν ευάλωτες καταστάσεις και σειράξει Και για αυτούς τους λόγους έλαβε τη δέσμευσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πλαίσιο των συνολικών δεσμεύσεών της να αντιμετωπιθεί ο στόχος του 0,15 έως 0,20 του ΑΕΠ που θα χορηγείται στην βοήθεια των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Αυτές οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν οι ίδιες την ευθύνη για την ίδια τους τη δική τους ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες ε, για να βοηθηθούν αυτές οι χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση αυτών των διαδικασιών ε, για την χρηστή ε, καλή διακυβέρνηση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, σωστή ε, διαχείριση. Είμαστε πεισμένοι εν τέλει ότι όλες οι χώρες έχουν την ευθύνη να βοηθήσουν τις φτωχότερες χώρες να ξεφύγουν από την παγίδα της φτώχειας και να μπορέσουν να σημειώσουν πρόοδο. Η πρόοδο σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες συνδέεται με τη συνεκτική μορφή και ε, συνάφεια της πολιτικής που θα ακολουθηθεί από τις προηγμένες χώρες που θα τις βοηθήσουν. Γι' αυτό η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών βοήθειας είναι σημαντική υπόθεση σε αρκετέ περιπτώσει ε, ζήτησε από άλλου χορηγού ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθούν σε αυτέ τι απαιτήσει. Οι αναδυόμενε ε, οικονομίε πρέπει και αυτέ να συνεισφέρουν στο μέτρο που του αρμόζει σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ θα λάβει τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πιο πριν από πλευρά Νικολάη ε, ε, υψώθηκε η ε, κιανή κάρτα, η μπλε κάρτα. Υποθέτω ότι θέλετε να παρέμβετε στο CASDI. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα για να θέσετε ερωτήσει ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε στο Συμβούλιο. Αυτό που θέλατε ήταν νομίζω να, να σας λάβω υπόψη εγώ ω πρόεδρος για τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στερότερα. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριο Φίλε, εξ ονόματο τη Επιτροπής. Να παρουσιάσει λοιπόν Λοιπόν τη δική του δήλωση. Παρακαλώ κύριε Φιούλη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για την επιτυχία της τέταρτης διάσκεψης των Εθνών για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη και κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια νέα ατμόσφαιρα δυναμική προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια, η πείνα και να τονωθεί η οικονομία στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Αυτή η δέσμευσή μας εκφράζεται μέσω των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και επίση εγκρίναμε κατευθυντήριε γραμμέ για τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην επικείμενη αυτή διάσκεψη για τι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Επίσης σημειώνουμε ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θα εκπροσωπηθεί πολύ δυναμικά μέσω τη αντιπροσωπείας του η οποία θα έρθει στην διάσκεψη. Πολλέ από τι λιγότερο ανεπτυγμένε αυτέ χώρε έχουν σημειώσει πρόοδο στην άπτυξή του. Η πρόοδος όμως ήταν άνηση και ακόμα πρέπει να γίνει πολύ σημαντική δουλειά. Λίγες μόνο από τις λιγότερο αντιγμένες χώρες ξεφεύγουν από την κατηγορία αυτή. Υπάρχουν πολλές άλλες οι οποίες οπισθοδρομούν ή αργούν πολύ όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Έτσι λοιπόν οι δωρητέ αλλά και οι ίδιε συναπτυσσόμενε χώρε θα πρέπει να διδαχθούν πολύ σημαντικά διδάγματα από τι επιτυχίε που έχουν πετύχει ορισμένε λιγότερο αναπτυγμένε χώρε, ιδίω μέσω τη εφαρμογή του προγράμματο των Βρυξελών. Η αμοιβαία ευθύνη και η παγκόσμια εταιρική σχέση είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία της διάσκεψης. Πρόκειται για μια κοινή πρόκληση. Οι εναπτυσσόμενες χώρες φέρουν πολύ σημαντική ευθύνη για τη δική τους την πρόοδο. Θα πρέπει να σχεδιάσουν και να ελοποιήσουν τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να πετύχουν τη χρηστή διακυβέρνηση. Όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός και επιτυχής εταίρος τους στην υλοποίηση των δεσμεύσεών τους, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, όσον αφορά τους κανόνες για την προέλευση και όσον αφορά την εξάλληψη του χρέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος δωρητής για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Τριπλασιάστηκε μάλλον η υποστήριξή μας προς τις χώρες αυτές κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη θα ζητήσουν και από άλλους εταίρους και από άλλες χώρες να κάνουν ανάλογες δεσμεύσεις με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δείξουν ανάλογη φιλοδοξία έχουμε την ευθύνη για την υποστήριξη των χωρών αυτών. Πρέπει να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ να βγουν από το καθεστώ φτώχεια. Επομένω, μια παγκόσμια εταιρική σχέση προ τι αναπτυσσόμενε χώρε, μάλλον και οι αναπτυσσόμενε χώρε, θα πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο τη ευθύνη του. Πρέπει να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ να σωματωθούν σε ένα κλίμα οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σημαντικό για αυτέ τι χώρε. Ο ιδιωτικό τομέα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί να επηρεάσει πολύ σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων, δημιουργώντας πλούτο και θέσεις εργασίας. Ε, δυναμική που έχει το εμπόριο προκειμένου να δημιουργήσει απασχόληση και να τονώσει την οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως υπογραμμίσει ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση όσον αφορά την πρόοδο και την ανάπτυξη και οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρες θα πρέπει να διέπονται και από δημοκρατία, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνη και χρηστή διακυβέρνηση. Η πρόοδο στις λιγότερο αναπτυγμένε χώρες συνδέεται με την ποιότητα και τη συνεκτικότητα των πολιτικών ανάπτυξη όλων των παγκοσμίων εταίρων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κατεβληθούν πολύ σημαντικέ προσπάθειε για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών υποστήριξη και βοήθεια και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική για την ανεπτυξιακή βοήθεια. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Προεδρία αναφέρθηκε ήδη σε τρει προτεραιότητε. Θα ήθελα εγώ απλώ να προσθέσω ότι η διάσκεψη θα πρέπει να ασχοληθεί και με το ζήτημα τη διαβάθμιση. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει ένα πιο αποτελεσματικό μηχανισμό προκειμένου να υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη προς τις χώρες αυτές που σιγά σιγά βαθμιαία βγαίνουν από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να περάσουν από την κατηγορία των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών σε μια καλύτερη κατάσταση την επόμενη δεκαετία. Σας ευχαριστώ. Εξ των πολιτικών ομάδων τώρα. Πρώτα για το Λαϊκό Κόμμα η κυρία Θεοχάρους για 1,5 λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε συνάρτηση με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από αποτελεσματικά μέτρα για να στηριχτεί η όλη προσπάθεια. Βεβαίω, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε θα είναι εξοπλισμένη και με ένα καλό ψήφισμα που εκφράζει, μπορεί που εκφράζει ικανοποιητικέ θέσει ωστόσο υπάρχει πρόβλημα με το στάτους της αντιπροσωπείας διότι ως παρατηρητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα για άμεση παρέμβαση και νομίζω ότι η επιτροπή και ο πρόεδρος μπαρόζο μπορούν να κάνουν μια, σημαντική παρέμβαση για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση διότι η ανάπτυξη και η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ένωσης και ο έλεγχος των μεταναστευτικών ρευμάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα δισεκατομμύριο περίπου πολίτες να ζουν στην αθλειότητα και στην φτώχεια φαίνεται ότι οι προσπάθειες για την ανάπτυξη των χωρών ε, των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών πρέπει να αναθεωρηθούν διότι φταίνουν βεβαίως και οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αλλά φαίνεται ότι δεν είναι και αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της φτώχειας. επισημαίνω ότι η εκμετάλλευση του πλούτου στις υποανάπτυκτες χώρες γίνεται από άλλους πλην των γηγενών πληθυσμών και ότι το δημοκρατικό έλλειμμα και η διαφθορά αλλά και η ανασφάλεια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των χωρών αυτών. όλα αυτά οδηγούν στην έλλειψη βασικών υποδομών στους τομείς της παιδείας της υγείας των συγκοινωνιών των επικοινωνιών της πρωτογενούς παραγωγής της γεωργίας του τραπεζικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης. νομίζω ότι στην κωνσταντινούπολη μπορεί να τεθούν οι μηχανισμοί για μια καλύτερη ε, προσπέλαση του φαινομένου της φτώχειας. ευχαριστώ. Για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Μπέρμαν για 1,5 λεπτό. Dank u, voorzitter. Een economische groei van 7%. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. <clears throat> Για αυτή την ανάπτυξη 7% οικονομική ανάπτυξη και περισσότερα παιδιά που θα πηγαίνουν σε ανώτερες σχολές και δημοκρατικά αιτήματα που διατυπώνονται στις λιγότερες ε, ε, χώρες είναι αυτό εφικτό και πρέπει εδώ να πει κανείς ότι σε σχέση με τα κονδύλια τα οποία ε, πρέπει να διατεθούν οι ε, χώρες, οι πλούσιες χώρες ε, με την διαγραφή χρέους μεριμνούν για να υπάρξει τέτοια ανάπτυξη. Αλλά δεν έχουμε φτάσει με κανένα τρόπο αρκετά μακριά. Δεν μπορεί αυτή η ανάπτυξη να διασφαλίσει αυτή την προοπτική και η φτώχεια εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη ανάγκη βλέπουμε ότι άνθρωποι ζουν με δύο δολάρια ε, ημερήσια αμοιβή και όλα αυτά δεν επαρκούν. Είναι παράλογο να λέει κανείς ότι η αναπτυξιακή πολιτική δεν λειτουργεί καθόλου. Έχουμε λίγες ευκαιρίες που δώσαμε και πρέπει να δοθούν περισσότερες. Η Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να καταλήξει στα αντίστοιχα συμπεράσματα και θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη κατανομή, καλύτερος επιμερισμός αγαθών και πλούτου. Έτσι θα μειωθούν οι εντάσεις. Κοινωνική ισότητα δίνει πολύ μεγαλύτερη ειρήνη από ότι οι ανισότητες των δικτατορικών καθεστώτων όπου μια ολιγαρχία και μια ελίτ πλουτίζει. Και εδώ πρόκειται να, για την δημιουργία δυνατοτήτων να επιτεθούν οι στόχοι για την ανάπτυξη και για τις οικογένειες και για την υγεία. Για μια φτωχή χώρα ε, ένα τέτοιο πρόβλημα ε, μπορεί να είναι πραγματικά ολέθριο. Πρέπει να βοηθήσουμε. Γι' αυτό πρέπει η δημόσια υγεία να χρηματοδοτηθεί και να διασφαλιστεί. Να διασφαλιστεί. Δεν πρόκειται μόνο για κονδύλια, αλλά πρόκειται και για νοσοκομεία και κλινικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το 1980 μέχρι το 2011 το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 19 3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετά μέσα για να εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια. Αυτά όσον αφορά την αριθμητική. Όσον αφορά την πολιτική, η βελτίωση τη μοίρα των πιο φτωχών δεν είναι τόσο προφανή. Πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητε επιλογέ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στοχεύσουμε τι πιο φτωχέ χώρε στα προγράμματα συνεργασία μα. Ε, και βεβαίω, κατά συνέπεια θα πρέπει να αποσυρθούμε σταδιακά από τι αναδυόμενε χώρε. Η Κίνα, ο πρώτο πιστωτής των ΗΠΑ, έχει αρκετά μέσα στη διάθεσή τη για να αντιμετωπίσει την φτώχεια εντό των συνόρων τη. Τρίτον, χρειάζονται ισχυρέ εταιρικέ σχέσει με τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Αυτέ θα κάνουν τα βασικά. Αλλά εμεί πρέπει να τι συνοδεύσουμε με, το, με την τεχνογνωσία μα, με την πραγματογνωμοσύνη μα, με την πολιτική μα βούληση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και τελευταίο σημείο, καθώ είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητέ, θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τη σωστή ηγετική θέση σε αυτή τη διάσκεψη. Mr. President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Θεοχάρους ε, αναφέρθηκε στο καθεστώς που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ε, διάσκεψης των μένων εθνών. Είμαστε ένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει πολύ γρήγορα να διευθετήσουμε το θέμα αυτό. Είμαστε όντως ο μεγαλύτερος δωρητής για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και όντως έχουμε βοηθήσει τα τελευταία χρόνια. παρόλα αυτά η φτώχεια δεν έχει μειωθεί. Πριν από δέκα χρόνια ο Πασκάλ Λαμή και η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, προχώρησαν στην πρωτοβουλία όλα εκτός από τα όπλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως το έκανε αυτό όλα εκτός από αγροκτήματα δεν έχουν βιομηχανική ικανότητα οι χώρε αυτέ, έχουν όμω τη δυνατότητα να πτυχθούν γεωργικά. Αν πραγματικά θέλουμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια, αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού, θα πρέπει να δυναμώσουμε τι ικανότητέ του να εμπορεύονται τα προϊόντα του. Δεν είναι η βοήθεια που θα μειώσει τη φτώχεια, αλλά το εμπόριο θα μειώσει τη φτώχεια. Προκειμένου να μειώσουμε τη φτώχεια και να αυξήσουμε το εμπόριο, θα πρέπει να επιτρέψουμε στι χώρε αυτέ να προχωρήσουν σε εξαγωγέ. Και οι χώρε αυτέ μπορούν να εξάγουν γεωργικά κυρίω προϊόντα. Προκειμένου όμω να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να εγκρίνουμε τις παράλληλες πολιτικές, τις κατάλληλες πολιτικές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι από τις 51 περίπου χώρες, τρεις μόνο κατάφεραν να ξεφύγουν από την κατηγορία των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός των ε, χωρών που δεν περιλαμβάνονται πλέον στην κατηγορία αυτή. κυρία για ένα λεπτό. Θα ήθελα ουσιαστικά τους δύο εκπροσώπους ε, Επιτροπής και Συμβουλίου να ρωτήσω γιατί πιστεύουν ότι σε αυτό το θέμα μπορούν με κάποια, κάποια στερεότυπα να αναφερθούν. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύνοδο της ε, Κωνσταντινούπολης, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπομισθούν επιτέλους πλήρως τις ευθύνες τους για την χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας και δεν μπορούμε να ανεχθούμε τα κράτη-μέλη αυτές τις ευθύνες να τις απεμπολούν όλο και περισσότερο. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι καθημερινά πεινούν και θα πρέπει οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, να δούμε ότι αυτές έχουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων που πεινούν. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτών των χωρών και αυτό το μέρος ε, να δούμε ότι το τμήμα το ε, έχει ακόμα πρέπει να μειωθεί. Για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους που πεινούν μιλάμε και ελπίζουμε ότι θα είναι πιο ανθεκτικές ε, όπως λέγεται οι λιγότερο ανεκτυγμένες χώρες. Αλλά κουραστήκαμε πλέον να ακούμε μόνο λόγια. Πρέπει συγκεκριμένες πράξεις να αναλυφθούν για να βοηθηθούν αυτές οι χώρες. Ευχαριστώ. Για τους μη εγγεγραμμένους ο κύριος Κλέης για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα αυτό. Πρόκειται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και σίγουρα είναι μια καλή ευκαιρία αυτή για να μιλήσουμε για το νόημα που έχει η αναπτυξιακή βοήθεια και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι ότι ε, οι περισσότεροι, όσο περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια υπάρχει τόσο ε, πιο ωραία ε, μπορεί να θεωρηθεί η κατάσταση. Βλέπουμε ότι σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια διατηρούνται μόνο μεγάλες γραφειοκρατικές δομές, η διαφθορά και η αυτοικανοποίηση των ε, αρχών στην ε, Αφρική. Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ανεξαρτησίας και πραγματικής ανεξαρτησίας. Η αναπτυξιακή βοήθεια δεν δίνει πολλά πράγματα όσο παράλογο και αν ακούγεται. Η αναπτυξιακή βοήθεια είναι μία από τις αφορμές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Αφρικής σήμερα. Πρέπει πραγματικά να βοηθήσουμε να αλλάξουμε πορεία, να αλλάξει αυτή η κατεύθυνση και να μην ε, δίνεται αυτή η βοήθεια μόνο στους ε, εξουσιαστές, σε αυτούς που έχουν την εξουσία, να μπορεί να φτάνει ως τους πολίτες, γιατί διαφορετικά σταματάς στη διαφθορά. Ευχαριστώ. Nou, Μπορείτε να δεχτείτε μια ερώτηση. Μάλιστα θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι εξωτερικά συμφέροντα ή συμφέροντα αλλοδαπών και άλλων χωρών στην Ευρώπη και στις, σε άλλες χώρες μερίμνησαν ώστε να παραμείνουν δικτατορικά καθεστώτα στην εξουσία και ότι αυτά σήμερα πλέον δεν λειτουργούν και ότι δεν ανελήφθη καμία προσπάθεια όσον αφορά τη σταθεροποίηση τέτοιων χωρών όπως στην Αφρική και αλλού. Λοιπόν, δημοκρατία αλλά και δημοκρατικά κινήματα. Αυτό σημαίνει εδώ πραγματικά αυθεντική δημοκρατία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αυθεντική σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια. Και θέλω να προσθέσω ότι εν μέρη συμφωνώ με αυτά τα οποία ο συνάδελφο Μπέρμαν προανέφερε. Πραγματικά εμεί ευθυνόμαστε διότι δικτατορικά καθεστώτα παρέμειναν στην εξουσία και μπόρεσαν να αγκιστρωθούν στην εξουσία. Με την Κούβα το είδαμε αυτό ανάγλυφα. Ο Φιντέλ Κάστρο ήταν ένα εταίρο, λέει με τον οποίο μπορούσε κανεί να συζητεί. Και αγκιστρώθηκε και αυτό στην εξουσία. Αυτό θα έπρεπε να ανήκει στο παρελθόν, να το έχουμε ξεπεράσει και πρέπει να μιλάμε για ανθρώπους που θα έχουν εκλεγεί δημοκρατικά με εκλογές και που θα έχουν με την εξουσία αλλά και που θα νοιάζονται για τους πολίτες τους και τη χώρα Σας ευχαριστώ πρόεδρε κυρίες και κύριοι οι ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, που η έννοια αυτή χρησιμοποιήθηκε για να ταυτοποιηθούν εκείνες οι κοινωνίες και κοινότητες που χρειάζονται τη μεγαλύτερη βοήθεια. Ο ορισμός αυτός βασίζεται όχι μόνο στο εισόδημα ανακεφαλή αλλά επίσης λαμβάνει υπόψη και άλλα στοιχεία όπως ε, το ανθρώπινο κεφάλαιο ως αναπτυξιακό παράγοντα. Είναι αξιοπερί, αξιοπρόσεκτο ότι οι περισσότερες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες βρίσκονται στην Αφρική. Αληθεύει λοιπόν, λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την Ήπειρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ότι ε, σε σχέση με τον αριθμό των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών αυτό αναπτύσσεται, αυξάνεται αυτό ο αριθμό. και μόνο τρει χώρε κατάφεραν να ξεφύγουν από την κατηγορία των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών. Γι' αυτό στη σύνοδο αυτή θα πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε πώ θα μπορέσουμε να καθορίσουμε μια στρατηγική για τι χώρε αυτέ που θα μπορέσουν να ε, ξεφύγουν από αυτή την κατηγορία με αποτελεσματικά μέτρα, με μια μια διαδικασία που θα είναι εύκολο να επιτηρηθεί. Χαίρομαι για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν μέτρα και προτάσεις για να βοηθηθεί αυτή η ε, εξέλιξη. Και inclusive growth, η συνολική σφαιρική ε, ανάπτυξη, μετρήσιμη ανάπτυξη είναι ένα τέτοιο στοιχείο. Η ανάπτυξη είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη ε, σημασία για την, την πρόοδο αυτών των χωρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι χρειαζόμαστε έναν απτό στόχο να αποφασιστεί στην συνάντηση της κωνσταντινούπολης και ο στόχος αυτός θα πρέπει να είναι να μειώσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στο μισό από ό,τι είναι σήμερα να μειωθεί ο αριθμός του στο μισό. Ακούγεται αυτονόητο κάτι τέτοιο, όμως εδώ και 30 χρόνια καταφέραμε, κατάφεραν αυτές οι χώρες, μόλις τρεις από αυτές τι χώρες να βγουν από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για να το πετύχουμε θα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας για να συμβάλλουμε κάθε χρονιά στο 0,15 με 0,20 του GNP μας για να έχει βοήθεια στις χώρες αυτές. Το ίδιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε τη συνοχή των πολιτικών μας για την ανάπτυξη policy coherence for development. Δεν μπορούμε από τη μία να δίνουμε χρήματα σε αυτές τις χώρες και από την άλλη στην ουσία να τους τα κλέβουμε μέσα από άδικες εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές πρέπει να πληρώσουμε το κλιματικό μα χρέο και αυτό σημαίνει επίση επένδυση σε αυτέ τι χώρε τόσο πολύ για την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή αλλά όσο και για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή αλλά και το χρέο μα το συσσωρευμένο χρέο μα από ε, τι αδικίε τη κοινή αγροτική μα πολιτική. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να προωθήσουμε την ε, διατροφική κυριαρχία, το food sovereignty αυτών των χωρών, προωθώντα παραδοσιακέ αγροτικέ πρακτικέ, τοπικού πόρου, τοπικέ καλλιέργειε και τοπικέ αγορέ και επίσης να αποτρέψουμε τις κερδοσκοπικές επιθέσεις την αρπαγή γης και τα μονοπόλια σπόρων που απειλούν όλους μας αλλά ιδιαίτερα ακόμα περισσότερο αυτές τις αδύναμες χώρες. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Αρσένη, ο κύριος Ντέβα έχει μία ερώτηση για σας. Τη δέχεστε. Mr. Deva, 30 seconds. I wonder whether my, the honorable... Αναρωτιέμαι αν ο αξιότιμος κύριος θα συμφωνήσει μαζί μου γιατί χρησιμοποίησε μια πολύ έντονη διατύπωση ότι κλέβουμε από τις αναπτυσσόμενε χώρε ότι για παράδειγμα δίνουμε 2 εκατομμύρια σε ένα μικρό ε, νησί για 70.000 τόνους, ε, ε, τόνου που πολλούνται στους δρόμους της Ευρώπης ε, για 23 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό κάνουμε με την ε, ε, αλληλευτική μας πολιτική. Και ο κύριος Δέβα, σε μεγάλο βαθμό οι αλληλευτικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες είναι ένα θέμα που χρήζει να επαναξεταστεί σε, σε βάθος είναι απαραίτητες είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή ένωση να είναι η χώρα που, αυτές, που συμφωνεί με αυτές τις χώρες έχει αυτή τη συμφωνία με αυτές τις χώρες και την πρόσβαση στα αλλιεύματα γιατί είναι η χώρα που το κάνει με τον πιο βιώσιμο δυνατό τρόπο όμω χρειάζεται να δούμε το πόσο πραγματικά τα χρήματα που δίνουμε σαν ανταλλάγμα για τα ψάρια και τα λιεύματα είναι επαρκή και πηγαίνουν σε αναπτυξιακή βοήθεια και βοηθάνε αυτέ τι χώρε τελικά να ορθοποδήσουν να βγουν από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Ευχαριστώ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι Λοιπόν, θα έλεγα ότι ο Υπουργό Νέμετ ναι, δεν έχει δίκιο σε σχέση με την κατάσταση των χωρών που ε, μπορούν να εκφύγουν από την κατηγορία των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών και ότι αυτό είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπαν ο κύριο Νίλ Ντέβα και ο κύριο Αρσένη. Τα τελευταία δέκα χρόνια μόνο τρει χώρε, η Μποτσουάνα, το πράσινο ακροτήριο Καμποβέρδε και οι Μαλδίβες ε, κατάφεραν να ξεφύγουν από αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή το κύριο αίτιο για αυτή την κατάσταση είναι η ε, ε, φτώχεια, έχουμε, η διαφθορά. Έχουμε χώρες που δεν έχουν φυσικούς πόρους. Για παράδειγμα την Ιαπωνία. Από την άλλη πλευρά έχουμε πλούσιες χώρες που έχουν πολλούς φυσικούς πόρους αλλά είναι πολύ φτωχές. Παράγει λοιπόν φτώχεια αυτή η παγίδα, αυτή η κατάσταση. Και ε, βλέπουμε ότι η συνδρομή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πέρα από την διάνοιξη νέων δυνατοτήτων πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί στην πολιτική συνδρομή να τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν σταθερές δημοκρατικές κυβερνήσεις να καταπολεμηθεί η διαφθόρα. Uh, Δέκα αιτήματα για τη δικασία Catch the Time. δυστυχώ έχουμε καθυστερήσει πολύ σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έξι μόνο μπορούν να πάρουν το λόγο. Ζητώ συγγνώμη από του άλλου τέσσερι. Αυτοί που θα μιλήσουν οι ακόλουθοι. Mr. Cortes Lastra, Ms. Stilla, Mr. Nicolai and Mr. Ferreira. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους που είχαν ζητήσει το λόγο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα είμαι πολύ αυστηρός με το χρόνο. Σας... ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι μια καλή ευκαιρία για να επανεξετάσουμε την διεθνή πολιτική αρρωγή για το εμπόριο. Αυτή η κατηγορία χωρών αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες για τις ε, οικονομικές ε, συναλλαγέ συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Η διαρκής αύξηση των τιμών των τροφίμων και μάλιστα ειδών πρώτης ανάγκης είναι τεράστιο πρόβλημα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ο κύριος στόχος αυτού του εμπορίου είναι η αύξηση, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας αυτών των 48 χωρών και εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να ξεριζωθεί η φτώχεια και να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά οικονομική βοήθεια ώστε να επιτεθούν οι στόχοι της χιλιετίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρε. Επίσης, η συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών πρέπει να εξεταστεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Μεταρρύθμιση δηλαδή των πλαισίων των εμπορικών σχέσεων. Κύριε Πρόεδρε, Βλέπουμε ότι η δική μας πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας έχει βοηθήσει τις χώρες αυτές να σημειώσουν πρόοδο. Βλέπουμε όμως και πως έχει κατηγοροποίηση των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τα μέσα και τις πολιτικές μας. Οι χώρες αυτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη φτώχεια και στις διενέξεις. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τρία ακόμα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε του εσωτερικού παράγοντε, όπω η διαφθορά, το ότι δεν η υπάρχουν απαραίτητε εγγυήσει για τη δημοκρατία, το ότι ε, δεν υπάρχουν απαραίτητοι παράγοντε προκειμένου να βοηθηθούν οι χώρε αυτέ. Σε οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την προσέγγιση μα, βοηθώντα περισσότερο τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, του γεωργού, καθώ επίση και την καλύτερη διαχείριση των πόρων του κράτου. Τέλο, θα πρέπει τα δικά μα μέσα ανεπτυξιακή βοήθεια να είναι καλύτερα στοχευμένα και να ε, συντονίζονται περισσότερο με την επιτόπου δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε με τι χώρε αυτέ, θα τονώσουμε τον ιδιωτικό τομέα και θα καταφέρουμε να τι βοηθήσουμε να βγουν από την κατηγορία αυτή για τα επόμενα δέκα χρόνια. Εδώ και δέκα χρόνια οι χορηγικέ χώροι συμφώνησαν για ένα πρόγραμμα δράσης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θεσπίστηκαν στόχοι για την αντιμετώπιση τη ε, ακραία φτώχεια σε αυτέ τι χώρε. Είναι προφανέ ότι οι λιγότερε ανεπτυγμένε χώρε είναι εκείνε που υφίστανται τα πλήγματα από την οικονομική κρίση όσον αφορά και το περιβάλλον και την αύξηση των τιμών ε, των ε, αγαθών. Δεν έχουμε όμω πετύχει αυτού του στόχου και μόνο δύο χώρε από τι 48 που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία κατάφεραν να μην είναι πια λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε. Βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Η επόμενη σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη θα επανεξετάσει το όσα έγιναν και θα ε, θεσπίσει ένα νέο πρόγραμμα δράση. Πρέπει να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μα για αυτέ τι χώρε και να πούμε ότι σε 10 χρόνια μάθαμε τα μαθήματα από την προηγούμενη ε, περίοδο και είμαστε σε θέση να παράσχουμε αποτελεσματική βοήθεια με τρόπο να υλοποιηθούν οι στόχοι μα. Όχι το 2020, αλλά το 2015, λαμβάνοντα υπόψη τι δεσμεύσει μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Συμβούλιο και την Κομισιόν και όλους όσοι μίλησαν. Υπάρχουν ε, κάποιοι ε, στόχοι που είναι ευπρόσδεκτοι σχετικά με τις ε, χώρες αυτές. Όμως θα κάνω μια ερώτηση. Η διατροφική ασφάλεια θα είναι μέρος των συζητήσεων αυτών. Στην υποσαχάρια Αφρική το 80% των αγροτών είναι γυναίκες. Αν, μπορέσουμε, αν μπορέσουν να εφαρμόσουν καλύτερες ε, γεωργικές μεθόδους, ε, αν επενδύσουμε σε τρόπους που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τον επιστημισμό των χωρών αυτών, θα είναι τεράστια η συμβολή μας. Εύχομαι ε, καλή επιτυχία στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, στην διάσκευση, αλλά επίσης θα περιμένω με ανυπομονησία τι θα έχουν να μας αναφέρουν αυτοί που θα παρευρεθούν εκεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είμαι πεισμένη Πρόεδρε ότι το Σώμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ένα κοινοβούλιο που είναι υπεύθυνο και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγχείρημα διεθνούς αλληλεγγύης στην καταπολέμηση της φτώχειας θα είναι κάτι που θα λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την χρήση των κονδυλίων που διατίθενται από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Έχουμε ευθύνη. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω ως ιδέα αυτή η διάσκεψη να αποτελεί για μας κίνητρο να εξετάσουμε το πρότυπο αλληλεγγύης που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα από πλευρά μας. Διότι αν εξετάσουμε αυτά τα οποία αποκαλούμε ως κατηγορία λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη, έχουμε φτωχές χώρες από τη μία πλευρά και άλλες χώρες που είναι πλουσιότερες. Πρέπει να επανεξετάσουμε λοιπόν την βοήθεια που δίνουμε και την αλληλεγγύη που εκφράζουμε. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό θα υπάρξει ο κίνδυνος που θα ελοχεύει αυτή η βοήθεια να μην είναι θετική για τις χώρες αποδέκτες. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτή τη συζήτηση κάνουμε λόγο για τις λιγότερο φτωχές ε, χώρες ε, και τις πιο ευάλωτες χώρες ε, του πλανήτη. Περίπου 50 χώρες πάνω κάτω που υφίστανται ακριβώς τις, τα χειρότερα πλήγματα και πρέπει εδώ να ληφθούν υπόψη από τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι μυρολατρικά αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυρολατρικό. Το αντίθετο συμβαίνει. Κάποιες από αυτές τις χώρες, αρκετές από αυτές είναι πολύ πλούσιες, πλούσιες σε φυσικούς πόρους όμως ε, δεν υπάρχει σωστό σύστημα οικονομικό και δικαιοσύνη ώστε σε παγκόσμια κλίμακα να μπορούν ε, να αντιμετωπίσουν ασυμμετρικές καταστάσεις ε, και τις ανισότητες. Είναι το αποτέλεσμα του ελεύθερου εμπορίου, της εκμετάλλευσης από το κεφάλαιο και τους φορολογικούς παραδείσους. Επίσης και λόγω των σειράξεων που υποδαβλίζονται για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Εδώ χρειάζεται μια αυθεντική συνεργασία και αλληλεγγύη και βοήθεια για την ανάπτυξη ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και να βοηθηθούν στην ανάπτυξή τους αυτέ οι χώρε. Ευχαριστώ. για λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, νομίζω ότι η ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση δείχνει ότι όλοι συμφωνούμε όσον αφορά τους στόχους. Αυτό φαίνεται και στο κοινό ε, ψήφισμα που υποβλήθηκε από τις ε, πολιτικές ομάδες. Βασικά θα ήθελα να αναφέρω τους εξής βασικούς στόχους, τους οποίους όλοι συμφωνούμε. Πρώτα απ' όλα ότι τα, η διάσκεψη θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο στόχος προφανώς είναι να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές ώστε να βγουν από το καθεστώς των ελάχιστων ανεπτυγμένων χωρών. Έχουμε ε, βήματα πρόοδου όσον αφορά την ελάφρυνση του χρέους, την πρόσβαση στην αγορά, ε, καθώς επίσης και ε, αναπτυξιακή βοήθεια προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η συνοχή των πολιτικών μας θα πρέπει να διαπνέει όλους τους τομείς υποστήριξης της, των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Καταπολέμηση της ε, φτώχειας και η προτεραιότητα θα πρέπει να έρθει, όπως είπε πολύ σωστά ε, ο κύριος Στήλε, ε, στην, η στην επιστημιστική ασφάλεια, στη γεωργία και στις υποδομές. Και βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Ντεβά, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στο εμπόριο που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όλοι έχουμε αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρωταρχική ευθύνη των λιγότερων πνιγμένων χωρών για τη δική τους ανάπτυξη. Χρειάζεται, χρειάζονται ένα πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα και καλή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα, που είναι απαραίτητα για να αυξηθούν οι χώροι, οι πόροι τους. Τέλος, έστω και αν δεν έχουν πρακτικά καμία ευθύνη για την αλλαγή του κλίματο, οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε θα πληγούν περισσότερο από όλε τι άλλες. Και γι' αυτό έχουμε μια υποχρέωση να τι βοηθήσουμε να προσαρμοστούν σε αυτή την αλλαγή. Ε, καταλήγοντας, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε υποστήριξε ε, θερμά ε, το θέμα αυτό τη βοήθεια προ τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Νέμεθ για πέντε λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο. Κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το συνολικό ε, όγκο για τις ε, χώρες αυτές. Από τότε που θεσπίστηκαν το 2002 στην διάσκεψη του Μόντρεαλ οι υποχρεώσεις το Συμβούλιο επανέλαβε την ανάγκη να κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές που θα μπορέσουν να αντληθούν για αυτή την βοήθεια, εγχώριες πηγές για τους νέους καινοτόμους μηχανισμούς και υποστήριξη των ανεπτυγμένων κρατών από τον ιδιωτικό της, ε, τον ιδιωτικό τομέα και τις αναδιόμενες επιχειρήσεις και στη συνέχεια το Συμβούλιο επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σοβαρά να εξετάσει προτάσεις για καινοτόμου μηχανισμούς χρηματοδότησης με δυνατότητα δημιουργίας πλούτου και εισοδήματος με προβλέψιμη ανάπτυξη όσον αφορά των πιο φτωχών αυτών χωρών με δυνατότητα να σημειώσουν πρόοδο. Θα ήθελα Τούτων λεχθέντων να προσθέσω κι εγώ τα σχόλιά μου στην άποψη του Επιτρόπου Φίλε για το ότι είναι σημαντικό να έρθουμε στο ύψος των ε, δεσμεύσεων και υποχρεώσεών μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ επίσης με τα σχόλια που έκανε για το να αυξηθεί η σημασία εμπορίου μεταξύ λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλαβα έξι για την παράτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στι 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δηλώσει